Ladies and gentlemen, please be seated. We start. Καθίστε παρακαλώ για να ξεκινήσουμε. Come in, please. would like to welcome you to the joint... Uh, Σας καλωσορίζω λοιπόν στην κοινή συνεδρίαση ΣΕΝΤΕ και ΜΠΑΛΤΖ, Επιτροπή Ασφάλειας Άμυνας και Προϋπολογισμό για τη χρηματοδότηση της κοινή πολιτικής ασφάλειας και άμυνας. Είναι η δεύτερη συζήτηση που κάνουμε της έκθεσης. Συν εισηγητές είναι ο κύριος Έντβαρτ Κούκαν από πλευράς της Επιτροπής μας και ο κύριος Ταράντ της Επιτροπής Προϋπολογισμών Καλωσορίζω και τον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής Προϋπολογισμών και του δίνω λοιπόν το λόγο για να μας κάνει την ε, εισαγωγική παρουσίαση. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε και εκ μέρους της Επιτροπής Προϋπολογισμών θέλω να ευχαριστήσω τους δύο συνσηγητές, τον κύριο Κούκαν και τον κύριο Ταράντ για την εργασία που έχουν κάνει από την αρχή αυτής της διαδικασίας και τώρα που έχουμε 130 τροπολογίες. Είναι εκείνη η έκθεση με βάση το άρθρο 55 και θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και για την πολύ ειλικρινή και καλή συνεργασία ακόμη πριν ε, συντάξω το σχέδιο έκθεσης όταν εκπροσωπούσα την Επιτροπή Προϋπολογισμών στη διάσκεψη Προέδρων Επιτροπών είχαμε πει ότι είναι σημαντικό αυτό το θέμα και για τις δύο επιτροπές μας και θέλουμε η έκθεση αυτή να αναλυφθεί ως κοινό εγχείρημα. Φυσικά η χρηματοδότηση της κοινή πολιτικής ε, ασφάλειας και άμυνας είναι αναγκαία, είναι προφανές αυτό. Οπότε θα πρότεινα τώρα να συνεχίσουμε τη συζήτηση για την έκθεση και τις τροπολογίες. Ευχαριστώ πολύ λέει και η κυρία Φώτηγα. Και τώρα να δώσω το λόγο στον κύριο Έντβαρτ Κούκαν. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, κύριε κύριο Χούκαν. Καλησπέρα συνάδελφοι. Δεν θα με γιατί το σχέδιο έκθεσης το έχουμε ήδη συζητήσει δύο φορές στην Επιτροπή μας. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να επανέλθουμε. Να ασχοληθώ με τις τροπολογίες και τους συμβασμούς, ούτως ώστε να προωθηθεί η διαδικασία έγκρισης του ψηφίσματος. Καταρχάς, θέλω να ευχαριστήσω τα μέλη και των δύο επιτροπών που υπέβαλαν τροπολογίες Όπως είπε και ο αντιπρόεδρος της Επιτροπής που φιλοξενούμε εδώ, είχαμε 130 τροπολογίες. Δεν είναι ναι, και λίγες, αλλά είναι σημαντική η έκθεσή μας. Οπότε, τονίζω ότι στόχος μας είναι να βελτιώσουμε την έκθεση. Θα υποστηρίξω λοιπόν όλες τις τροπολογίες που συμβαδίζουν με το πνεύμα της έκθεσης. Τώρα για συμβαστικές τροπολογίες. Συνεδριάσαμε εισηγητές και σκιώδεις νωρίς σήμερα το πρωί και συμφωνήσαμε σε πέντε συμβαστικά κείμενα που καλύπτουν θέματα όπως η γενική χρηματοδότηση των αποστολών και της λειτουργίας στην παράγραφο 1 η πρόταση της Επιτροπής για χρηματοδοτικούς κανόνες, ο μηχανισμός Αθηνά και η χρηματοδότηση των στρατιωτικών επιχειρήσεων, παράγραφος 15 και 16. Να κάνω μερικές επιμέρους παρατηρήσεις. Ορισμένες παράγραφοι όπου θα ήθελα να διατηρήσω την αρχική κατευθυντήρια γραμμή της ε, έκθεσης. Στο 7, για παράδειγμα, θεωρούμε ότι πρέπει να συμπεριληφθεί το κέντρο κοινών υπηρεσιών καθώς ε, και οι αποθήκες του CSDP. Επίσης, η πρόταση στην παράγραφο 6 για να έχουν τη συνολική ευθύνη και για τα στρατιωτικά και μη στρατιωτικά θέματα οι στρατιωτικοί διοικητέ, θέλω να διατηρηθεί. Συμφωνώ με τι περισσότερε προτάσει που ασχολούνται για το τμήμα της συνέπειας και συμπληρωματικότητα. Αυτό αφορά ιδιαίτερα την ολοκληρωμένη προσέγγιση για την CSDP και την συνεργασία μεταξύ στρατιωτικών και πολιτικών αρχών. Το τμήμα τώρα για τη χρηματοδότηση των στρατιωτικών επιχειρήσεων. Όπως είπα, προσπαθήσαμε να έχουμε δύο συμβαστικές τροπολογίες για παραγράφους 15 και 16. Οι τροπολογίες αυτές ενημερώνουν την τελευταία απόφαση που λήφθηκε στο Συμβούλιο για το μηχανισμό Αθηνά. Για τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας έχουμε διάφορες τροπολογίες που θέλω να εξετάσω, ούτω ώστε να τις εντάξω σε ένα συμβαστικό κείμενο. Αυτό δεν μπόρεσα να το κάνω, λόγω των διαφορετικών απόψεων για το πώς θα μπουν στον προϋπολογισμό πιστώσεις για προσωπικό και τα τρέχοντα έξοδα του φορέα αυτού. Όπως ήδη αναφέρθηκε στην έκθεσή μας του 2012, όπως αναφέρθηκε λοιπόν σε αυτή την έκθεση. Οπότε θα υποστηρίξω όσες τροπολογίες πηγαίνουν προ αυτή την κατεύθυνση. Κάτι γενικό που θα ήθελα παρακαλώ να το λάβετε υπόψη σας στο τελικό κείμενο του ψηφίσματος Αυτά είναι κατά την άποψή μου τα πιο σημαντικά σημεία για τα θέματα που αφορούν τον συγκεκριμένο προϋπολογισμό θέλω παρακαλώ να ακούσω σχόλια και από τους συναδέλφους της Επιτροπής Προϋπολογισμών ευχαριστώ, αυτά είναι τα εισαγωγικά μου σχόλια Ευχαριστούμε κύριο Τάραντ Θα προχωρήσουμε στους κοιόδους εισηγητές, ε, γιατί δεν έχει φτάσει ακόμα ο κύριος Τάραντ. Η κυρία Γετεμάκη, Ανέλη Γετεμάκη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους ε, εισηγητές. Ε, είναι πολύ συνενετικός ο τρόπος που καθοδηγούν τη διαδικασία και σέβονται απόλυτα όλους τους συναδέλφους. Χαίρομαι επίσης ε, διότι υπάρχει μεγάλη σύγκληση σε απόψεις των πολιτικών ομάδων σε σχέση με τη χρηματοδότηση της κοινή ε, πολιτικής ασφάλειας και άμυνας. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τους ε, υπόλοιπους σκιώδεις εισηγητές, διότι είναι πολύ συγκεκριμένοι και, διεξο... και λεπτομερής η συμβολή τους στη διαδικασία. φαίνεται ότι η χρηματοδότηση της πολιτικής θεωρείται ότι προς το παρόν ε, παίρνει υπερβολικά πολύ χρόνο, δεν είναι αποτελεσματική, αυτό πιστεύουν όλες οι πολιτικές ομάδες και ε, αυτό που εις βάρος των αποστολών και επιχειρήσεων. Η αποτελεσματικότητα είναι η βασική στόχη για να έχουν μακροπρόθεσμα επιτυχία οι επιχειρήσεις της κοινή πολιτικής ασφαλείας και άμυνας. Ο μηχανισμός Αθήνα για τη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων ε, χρήζει ε, ριζικής μεταρρύθμισης Οι χώρες που συμμετέχουν στις επιχειρήσεις ε, καλύπτουν το μεγαλύτερο κόστος σε σχέση με αυτό που καλύπτουν οι ομολογοί τους ε, και αυτό θα πρέπει να ληφθεί υπόψη λόγω του υψηλού κόστους των επιχειρήσεων. Επίσης, χρειαζόμαστε καλύτερο επιμερισμό των ευθυνών βάσει της αξιολόγησης των επιπτώσεων κάθε αποστολής. Η χώρα μου, σε απόλυτους όρους, είναι από τις πιο δραστήριες χώρες που συμμετέχουν σε αυτές τις επιχειρήσεις. παρότι ε, έπληξε και τη χώρα μου σε μεγάλο βαθμό η χρηματοοικονομική κρίση, συμβάλαμε ε, σε μεγάλο βαθμό στη χρηματοδότηση. Και ελπίζουμε ότι εφ' εξής ε, θα έχουμε μια καλύτερη βάση για να συνεχίσουμε τις συζητήσεις για τη χρηματοδότηση. Ευχαριστούμε πολύ κυρία Φωτίγκα. Έχει έρθει ο κύριος Τάραντ, πλέον θέλετε το λόγο βεβαίως. Ε, διότι θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους που δείχνουν τόσο μεγάλο ενδιαφέρον για την έκθεση και για τις πολυάριθμες ε, τροπολογίες που έχουν κατατεθεί. Χαίρομαι πάρα πολύ ε, για τη συνεργασία, την αγαστή συνεργασία που έχουμε με τον κύριο Κούκαν και για να είμαι ειλικρινής ε, θα πρέπει να ευχαριστήσω και τον ε, κύριο Γκυγιόμ Μπλεγερ από... και όλους όσους συνεργάστηκαν μαζί μας από τις διάφορες επιτροπές. Είναι μεγάλες οι προκλήσεις και μεγάλες οι δυσκολίες που αντιμετωπίζει η κοινή πολιτική ασφάλειας και άμυνας και θα θέλαμε να έχουμε μια πιο φιλόδοξη πολιτική σε σχέση με τώρα. Επίσης, για να υλοποιηθεί αυτός ο στόχος, είμαστε διατεθειμένοι να προσφέρουμε και τα επαιτούμενα μέσα. Αυτό απηχείται στις τροπολογίες μας για τον μηχανισμό Αθηνά. Ε, βλέπουμε ότι ε, έχει αλλάξει η κατάσταση στο Συμβούλιο, έχει καταλήξει το Συμβούλιο σε μία συμφωνία όχι τόσο φιλόδοξη όσο ε, αυτή που ζητούσαμε εμείς μέσα στην έκθεσή μας. Σίγουρα δεν μπορούμε πλέον να απευθύνουμε την ίδια επίκριση στο Συμβούλιο ότι δεν καταλήγει σε συμφωνία. Εγώ στο μέλλον ε, θα κατηγορήσω το Συμβούλιο ότι δεν κατέληξε στην απαιτούμενη συμφωνία. Κάποια μέλη της Επιτροπής δεν έχουν καταθέσει τροπολογίες για τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας και κυρίως για την ένταξή του ε, στον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι ανακύπτουν πολλά ζητήματα Δεν έχει ζητηθεί όμως αυτό το θέμα ε, διεξοδικά στην Επιτροπή Προϋπολογισμών ε, από τα μέλη που ασχολούνται με τους οργανισμούς, από τα μέλη της Επιτροπής, βουλευτές δηλαδή που ασχολούνται με τους οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ίσως να χρειαστεί ξεχωριστή ψηφοφορία για τις ε, σχετικές τροπολογίες αν δεν καταλήξουμε σε συνένεση. Ε, τώρα για τις πολιτικού χαρακτήρα επιχειρήσεις εδώ και 10 χρόνια υπάρχει το ίδιο πρόβλημα με αυτές τις επιχειρήσεις και κατά τη σύνταξη της έκθεσης ήρθαμε σε επαφή με τον κύριο Κούκαν με την υπηρεσία εξωτερικής δράσης ακριβώς για αυτό το ζήτημα και καθώς και με τις αντιπροσωπείες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε διάφορες χώρες και καταλήξαμε σε μια αποδεκτή λύση η οποία όμως προϋποθέτει ότι θα ε, υιοθετήσουμε μια πιο φιλόδοξη προσέγγιση στην έκθεση. Δεν πιστεύω ότι είναι σκόπιμο να αποδυναμώσουμε το κείμενο, κυρίως θα μιλάμε για το κοινό κέντρο επιχειρήσεων. Το κέντρο κοινών υπηρεσιών, μάλλον. Ε, σας ευχαριστώ. Δεν έχω τίποτα άλλο να προσθέσω. Ευχαριστώ, λέει η κυρία Φωτίγα. Θα ήθελα να ακούσουμε τον κύριο Μπρούκ ε, από την ε, ΓΑΜΑ ΔΕΛΤΑ ε, προϋπολογισμού της Επιτροπής. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα είμαι πολύ σύντομο Από πλευράς Κομισιόν θα θέλαμε να επιστήσουμε την προσοχή σας στις τροπολογίες της Επιτροπής Προϋπολογισμών και στις τροπολογίες του Πρόεδρου και του κύριου Γκάγερ. Χαιρόμαστε που παρατηρούμε ότι μεταξύ των τροπολογιών της Επιτροπής αυτής έχουμε την παγιωμένη προσέγγιση για τους κανόνες ε, περί αποστολών στο πλαίσιο της CSDP είμαστε ικανοποιημένοι με αυτή την αλλαγή Α, ανησυχεί το ότι ζητάει η Επιτροπή εκχώρηση ε, των εξουσιών στον διοικητή το οποίο δεν είναι δυνατόν θέλουμε λοιπόν να στενεί τένο συντονισμό μεταξύ Επιτροπή και Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερική Δράση και στο άρθρο 61 καλούμε, γίνεται έκκληση για μια πλατφόρμα υποστήριξη που είναι το ίδιο με την υπηρεσία που υπάρχει, απλά μια εξέλιξη και για την τροπολογία 63. Θα θέλαμε επίση να υποστηρίξουμε το ζήτημα της συμπληρωματικότητας μεταξύ της ε, κοινή πολιτική ασφαλείας και άμυνας και των λοιπόν προγραμμάτων της ε, ε, Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης για την τροπολογία 117 του κ. Γκάιερ. Θα θέλαμε να διατηρηθεί μια γενική γραμμή για τις αποστολές πέραν των άλλων αποστολών που έχουν δει και του στον προπολογισμό. Γιατί αυτό δίνει την ευελιξία να μπορεί να στήσει κανεί εύκολα μια αποστολή κατά τη διάρκεια του έτου όταν καθίσταται απαραίτητο. Ευχαριστώ. Thank you, sir. Ευχαριστούμε. Ζήτω συγγνώμη. Ήταν δικό μου το λάθος ε, συγκεκριμένα. Δεν είδα την κυρία Λέζινγκ που είναι σκέωδης της ΓΚΟΕ. Έχετε το λόγο κυρία Λέζινγκ. Μικρόφωνο, μικρόφωνο παρακαλώ. Λοιπόν, με συγχωρείτε, ε, γιατί δεν ήξερα εάν όλοι οι σκιώδεις έπρεπε να πάρουν το λόγο τώρα αυτόματα. Γι' αυτό δεν ζήτησα το λόγο. Περίμενα όπως το σχολείο να μου πούν να, να πω την άποψή μου. Ποια είναι σύντομα η άποψη της ομάδας μου για την έκθεση. Θα μπορούσατε να φανταστείτε ότι έχουμε σοβαρές αμφιβολίες για τη βασική φιλοσοφία αυτής της έκθεσης. Ο στόχος ήδη έχει διατυπωθεί να είναι δυνατόν να χρηματοδοτηθεί όσο το δυνατόν περισσότερο η ανάπτυξη των δραστηριοτήτων άμυνας και ασφάλειας και της βιομηχανικής και τεχνολογικής βάσης για θέματα άμυνας ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα έχουμε συζητήσει επανειλημμένα τα θέματα αυτά και πάντα έχω πει σαφέστατα την άποψη της ομάδας μας ότι δηλαδή θεωρούμε ότι ερμηνεύουμε το άρθρο 142 η οποία ερμηνεία έχει επιβεβαιωθεί από πολλούς και όχι από τα μέλη της Επιτροπής ότι οι δραστηριότητες με στρατιωτικούς ε, στόχους δεν πρέπει να χρηματοδοτούνται από τον προπολογισμό της Ένωσης. Και τώρα η προσπάθεια αυτής της έκθεσης θεωρώ ότι προσπαθεί να βρει τρόπους να αποφύγει αυτό το άρθρο. Να μην αναφερθώ τώρα σε όλες τις λεπτομέρειες. Όλα αυτά που λένε για τη συνεργασία και την ε, βελτίωση της συνεργασίας και όλα αυτά. Ένα μόνο να καταστήσω σαφές. Ότι η στρατιωτική έρευνα δεν πρέπει να χρηματοδοτείται από τον ενησιακό προπολογισμό και ιδιαίτερα η έρευνα για να αναπτύξουμε τηλεκατευθυνόμενα αεροπλάνα drone της Ένωσης σε συνεργασία με τον Οργανισμό Ευρωπαϊκής Άμυνας. Τα απορρίπτουμε όλα αυτά για την επέκταση του μηχανισμού Αθηνά. Δεν θα αναφερθώ στα οικονομικά προβλήματα. Οι μικρές χώρες, οι οικονομικές αδύναμα, οι οικονομικά αδύναμες χώρες δεν μπορούν να συμμετάσχουν. Το βασικό για μένα είναι να υπάρχει η δυνατότητα δημοκρατικού ελέγχου που τώρα αποκλείεται. και με αυτόν τον τρόπο δεν πληρώνουν όλοι για το κόστος ανάλογα με το πώς το προκαλούν. Γιατί όλοι πρέπει να συμμετέχουν σε αυτό το μηχανισμό. Αν γίνει κάτι τέτοιο, οι κοινοβουλευτικές αρχές δεν μπορούν να εκφραστούν και να ελέγξουν. Δεν βλέπω πουθενά να γίνεται κάποια προσπάθεια να υπάρχει κοινοβουλευτικός έλεγχος από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Οπότε καταλήγοντας, υπάρχουν πολλοί λόγοι, τους οποίους ε, απλώς και αγράφησα, για τους οποίους απορρίπτουμε αυτή την έκθεση, θα υποβάλουμε μία έκθεση μειονότητας, μειοψηφίας. Πρόεδρος. Ναι, φυσικά ε, θα ήθελα να ε, δώσω το λόγο σε όλους τους σκιώδεις. Κύριε Φουνζουλίτσα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Αφού παρενέβησαν όλοι οι σκιώδεις είναι καθήκον μου φαίνεται να πάρω και εγώ το λόγο. Με μεγάλη ευχαρίστηση θέλω να επενέσω το έργο των δύο συγητών. Η εκθέση αυτή είναι εξαιρετική. Σήμερα το πρωί είχαμε μια συνάντηση μαζί τους για τις συμβαστικές τροπολογίες. Η συζήτηση υπήρξε επικοδομητική Φυσικά πέραν των τροπολογιών που υπέβαλα εγώ και ορισμένες από τις οποίες συμπεριλήφθησαν σε αυτές τις συμβαστικέ τροπολογίες θα υποβάλω φυσικά και τις υπόλοιπες τροπολογίες. Ουσιαστικά έχουν συμπεριληφθεί σε αυτή τη λίστα τροπολογιών. Συζητήσαμε λίγο για τη συμβιβαστική 5 στην παραγραφό 16 και εκεί είχα μια πρόταση να μην αντικατασταθεί η λέξη should με has to consider ε, καθώς μιλάμε για τη χρηματοδότηση των αποστολών αυτών και μετά ανταλλάξαμε απόψεις με τους δύο συγγητές και τους συναδέλφους μου και αποφασίσαμε ότι θα έχουμε μια προφορική τροπολογία επί της έκθεσης όσον αφορά την επίβλεψη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου επί του τρόπου με τον οποίο οι διάφορες αποστολές και επιχειρήσεις χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο της κοινή πολιτικής άμυνας και ασφάλειας. Αυτά θα παρουσιαστούν όλα εν ευθέτω χρόνο στους συναδέλφους και θα δούμε ποια θα είναι τα αποτελέσματα. Για άλλη μια φορά τα συγχαρητήριά μου στους δύο εισηγητές. Ευχαριστώ. Thank you. Ευχαριστούμε ο κύριος Άλλη. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Ήθελα και εγώ να αναφέρω ότι οι συγκεκριτές έκαναν εξαιρετική δουλειά. Τα καταφέραν πολύ καλά και με τις συμβαστικέ ε, για τα σημαντικά σημεία. Είναι επίκαιρη αυτή η συζήτηση, πρέπει να πω. Με αυτή τη συζήτηση και με αυτή την ε, έκθεση που έχουμε μπροστά μας, ε, τι πρέπει όμως να πετύχουμε. Πιστεύω το σημαντικότερο είναι ότι πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να αυξήσουμε τους προπολογισμού των κρατών μελών τη Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και όχι να πέσουμε κάτω από το 2% του ΕΕΠ ε, των χωρών, διότι με αυτό στο νου μας ε, πρέπει να επικεντρωθούμε περισσότερο στη συγκέντρωση ε, ικανοτήτων και στην κοινή χρήση δυναμικού και να διασφαλίσουμε την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα ώστε να εξοικονομήσουμε κόστος. Δεδομένης της απόφασης του ΝΑΤΟ για το ελάχιστο ποσό του 2% του ΕΕΠ ε, για τους προπολογισμούς των κρατών μελών ε, του ΝΑΤΟ και δεδομένης και της δήλωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι είπε ότι καλωσορίζει αυτή την απόφαση. Προς τα εκεί πρέπει να κινηθούμε και εμεί, και όπω είπε ο κ. Στεράν θα γίνουν συζητήσεις όσον αφορά ε, το συμβιβασμό για τον προπολογισμό τη Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Άμυνα, κατά πόσο θα συμπεριληφθεί στο κονδύλιο του Ευρωπαϊκού ε, Προπολογισμού ή αν θα αφήσουμε την κατάσταση όσο έχει αυτή τη στιγμή. Όπως ανέφεραν και οι λοιποί συνάδελφοι, ο μηχανισμός Αθηνά στα περισσότερα κράτη-μέλη δεν λειτουργεί όπως θα θέλαμε. Δεδομένου αυτού λοιπόν μπορούμε να παρατείνουμε τις συζητήσεις και να δούμε πώς θα προχωρήσουμε. Η συζήτηση αυτή λοιπόν πιστεύω που γίνεται στην εκθέση είναι πολύ επίκαιρη και υπάρχουν αρκετέ τροπολογίε που καθιστούν το θέμα εξαιρετικά ενδιαφέρον, αναγκαίο και επίκαιρο. Ευχαριστώ. Mr. Ευχαριστούμε κύριε Κάλβερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δεν θα σας εκπλήξει ούτε σας εδώ στην Επιτροπή, ούτε στη δική μου περιφέρεια, στο West Midlands, όταν θα πω ότι ναι, καλωσορίζουμε την ε, συνεργασία μεταξύ ε, κρατών μαλλών. Έχουμε ήδη όμως δομές όπως το ΝΑΤΟ και την ε, Οργάνωση για τη Συνεργασία και την Ασφαλεία στην Ευρώπη που ενθαρρύνουν τη συνεργασία όταν είναι αμοιβέ αποφελής. Ωστόσο, έχω και αμφιβολίες για τη συγκέντρωση αυτή της κοινή πολιτικής άμυνας και ασφάλειας και τη χρηματοδότηση με τον τρόπο αυτό. Ειδικότερα θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας στο μηχανισμό Αθηνά για, για την κοινή χρηματοδότηση των στρατιωτικών επιχειρήσεων. Το τρέχον ψήφισμα προβλέπει αύξηση του κόστους ε, και πολλές τροπολογίες ε, κάνουν έκκληση για αύξηση του, ε, των δαπανών για το μηχανισμό αυτό για ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Είναι απαράδεκτο όταν τα μεγάλα κόμματα του Ηνωμένου Βασιλείου αρνούνται να διατηρήσουν τις δαπάνες στο ελάχιστο του 2% παρότι αναμένουμε να αυξήσουμε τις δαπάνες ε, σε πολιτικές επιχειρήσεις. Είναι ε, σημαντικό κάθε κράτος μέλος να κρατήσει ευθύνες και ε, να αποφασίζει το ίδιο για τις δυνατότητες που θα προσφέρει ώστε να παρέχει τις... Να ζητήσω τώρα και από τους δύο συνεισηγητές να απαντήσουν στις ερωτήσεις και να μας πούν τα τελικά του σχόλια. Ο κύριος Κούκαν. Ευχαριστώ. Θα είμαι σύντομος. Ευχαριστώ όλους τους ομιλητές για τη συμβολή τους. Ευχαριστώ όσους ε, στηρίζουν τη βασική φιλοσοφία της έκθεσης. Μπορούμε φυσικά να συζητήσουμε τα επιμέρους Θέλω να είμαι σαφής. Καταλαβαίνω όσους υπέβαλαν τροπολογίες και συμπεριλαμβάνονται αυτά που τους ενδιαφέρουν στην έκθεση. Για την κυρία Λέζινγκ. Τι κατανοώ. Πλήρως. Κατανοώ τους λόγους που σας οδηγούν στην απόφαση να υποβάλλετε έκθεση μειοψηφίας. Το πρωί το συζητήσαμε το θέμα που έθεσε ο κύριος Φρουντζούλητσα. Μπορούμε να υποβάλουμε μια προφορική τροπολογία επί της οποίας θα συμφωνήσουν και οι υπόλοιποι συνάδελφοι. Ο κύριος Άλλη είπε ότι είναι πολύ επίκαιρη η συζήτηση του θέματος αυτού και διάφορα θέματα που πρέπει να διευκρινίσουμε πριν περάσουμε στην έγκριση της έκθεσης. Και τον κύριο Κάρβερ τον ευχαριστώ για την παρέμβασή του. Αυτά είχα να πω. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριο Σταράντ, λέει πρόεδρος. Συμφωνώ με τον κύριο Κούκαν. Α, ευχαριστώ πολύ, λέει πρόεδρος. Μα συμφωνούμε λοιπόν όλοι, περίπου. Άρα μπορούμε να κλείσουμε το θέμα αυτό. Η ψηφοφορία θα γίνει στην ΑΦΕΤ στις 14 Απριλίου. Ευχαριστώ τον Σύμπροεδρο και όλους τους συναδέλφους ε, που συμμετείχαν στη συζήτηση για την έκθεση. Σας ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ τα μέλη της ε, ΣΕΝΤΕ να μείνουν στην αίθουσα. Θα κάνουμε δύο λεπτά διακοπή και θα συνεχίσουμε αμέσως μετά με την έκθεση Γκόμες.